συνταχθούν. Σας ευχαριστώ πολύ πρώτον που συμμετείχατε στην ε, Ολομέλειας και όπως έλεγα, τα πρακτικά λοιπόν θα καταστούν, θα αποκληθούν ε, προ έγκριση στι αρχέ επόμενη Ολομέλεια ε, και αν δεν υπάρξει αντίρρηση, οι αποφάσει οι οποίε έλαβαμε σήμερα θα στους αρμόδιους φορές, αρμόδιες αρχές αρχέ.